the record. <laughs> off the record. buenos días, ahora ya en, en nuestra... Καλημέρα σας λοιπόν τώρα και από την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ε, δεχτήκατε να κάνουμε αυτή την αλλαγή, να τρέχουμε από τη μία αίθουσα στην άλλη και προχωράμε με την ημερήσια διάταξη. Ε, πρωτόκολλο σχετικά με τον καθαρισμό των αλληλευτικών δυνατοτήτων και τη χρηματική αντιπεροχή που προβλέπεται στη Συμφωνία Αλληλευτική Σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τη Δημοκρατία των Σεϊχελών. Σημείο 15. Ξέρετε σήμερα ότι θα συζητήσουμε ε, το θέμα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Πατράων Νέβε. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην συγγήτρια και μετά στην Κομισιόν, γιατί θα κάνουμε συζήτηση με την Κομισιόν. Κύριε Γκάλεχερ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι βλέπω, από τι εκκρεμότητε που έχουμε στην ημερήσια διάταξη και δεδομένου ότι είναι Πέμπτη και έχουμε και απογευματινή συνεδρίαση, θα ήθελα να προτείνω να συζητήσουμε τις συστάσει των συντονιστών σήμερα το πρωί, γιατί ίσω το απόγευμα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχουμε και κανέναν εδώ. Καλό θα ήταν να τα συζητήσουμε αυτά πριν από τι 12.30. Έχει κανεί αντίρρηση. Οι συστάσει είναι όντω το μόνο σημείο στο οποίο θα πρέπει να εγκρίνουμε κάποια απόφαση. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να σας πω απλώς ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και το γεγονός ότι είναι λίγοι οι συνάδελφοι που έρχονται εδώ στην Επιτροπή. Ε, πάντα βέβαια πληρώνω την ύφη αυτοί που, που είναι εδώ και όχι αυτοί που απουσιάζουν, αλλά ίσως στο τέλος θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ε, τα θέματα αυτά και το απόγευμα να κρατήσουμε την... Ε, ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο και την παρουσίαση της έκθεσης. Εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω το απόγευμα να έρχεται όσο το δυνατόν περισσότεροι. Κύριε Αρσένη, παρακαλώ. Όπως και εσείς κύριε Πρόεδρε, ανησυχώ λίγο γιατί δεν έχουμε και πολλούς συναδέλφους εδώ. Θα προτιμούσα λοιπόν να τηρήσουμε το πρόγραμμα και να συζητεί όπως ε, έχει προγραμματιστεί στην ημερήσια διάταξη και την ώρα που έχει αποφασιστεί να συζητηθεί. Ο κύριος Στίβενσον. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς εγώ δεν θα είμαι εδώ το απόγευμα. Πρέπει να φύγω για το Λονδίνο. Συμφωνώ λοιπόν με τον ε, Πάτε Κόπ. Ε, οι παρουσίες ε, μάλλον θα είναι λιγότερες το απόγευμα. Καλύτερα να το κάνουμε σήμερα το πρωί. Κοιτάξτε, εμεί δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για αυτούς που απουσιάζουν. Όσοι είναι εδώ είναι αυτοί που αποφασίζουν. Επομένως, έχουμε δύο προτάσεις να τις ψηφίσουμε όπως γίνεται συνήθως. Ή τροποποιούμε την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας ε, και μεταφέρουμε το σημείο στο, για το τέλος του πρωινό. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης του κυρίου Γκάλαχερ. Κατά δύο αποχές, καμία. Ωραία. Θα είναι το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης σήμερα το πρωί. Κύριε Πατράντα έχετε το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο σημείο λοιπόν που έχουμε δώσει στην ημερήσια διάταξη είναι η Συμφωνία Οικονομικής ε, Σχέσης ε, για τις ελευτικές δυνατότητες και τις χρηματικές αντιπεροχές που προβλέπονται στη Συμφωνία Ελευτικής Σύμπρακτης μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Δημοκρατίας των ΣΥΧΕΛΟΝ για τις Σεϊχέλες, η Αλία και ο τουρισμός είναι οι δύο βασικές ε, οικονομικές δραστηριότητες και θα πρέπει να τονίσουμε και το εξής. Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ε, τα έσοδα από την Αλία έχουν υπερβεί όλα τα έσοδα του τουρισμού. Να σας το εξηγήσω, για... μάλλον σας το εξηγώ αυτό για να σας πω ότι οι Σεϊχέλες παραδοσιακά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτή τη συμφωνία. Τους ενδιαφέρει επίσης ε, ε, και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης τους αλλοί στο θέμα αυτό. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να αναφερθούμε όμως και στο θέμα της πειρατείας. Eh, στην ε, πειρατεία η οποία δυστυχώς εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή και αυτό σημαίνει ότι κάποια σκάφη έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή και δεν αλλιεύουν εκεί. Η πειρατεία λοιπόν έχει συνέπειες. Ε, υπάρχουν κάποιες προβλέψεις που λένε ότι ίσως η, ε, η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχύσει λίγο το θέμα αυτό και επειδή ακριβώς είναι τόσο αντίξεως οι συνθήκες εξακολουθούν να υπάρχουν συμφέροντα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. από αυτά που σας εξήγησα μπορεί ε, λόγω των συνθήκων που επικρατών ε, να ε, εγκαταλείψουν την Αλία κάποια σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και η αλία τόνου στην περιοχή, αλλά οι τόνοι που βρίσκονται στην περιοχή είναι άκρως μεταναστευτικά είδη. Είναι ο τόνος του Ινδικού ωκεανού και σύμφωνα με την Περιφερειακή Οργάνωση Αλίας, τα αλλιεύματα τόνου στην περιοχή είναι πολύ χαμηλότερα από τις δυνατότητες που υπάρχουν, επομένως δεν υπάρχουν προβλήματα ε, όσον αφορά τη βιωσιμότητα για τη συγκεκριμένη αλία. Τώρα, για τα πιο τυπικά του πρωτοκόλου, ισχύει για έξι χρόνια, θα υποκαταστήσει την προηγούμενη συμφωνία η οποία εξέπνευσε στις 17 Ιανουαρίου του 2014 και πρέπει τώρα να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε στις παρούσες συνθήκες ε, για την αλία στην περιοχή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώνουμε ότι έχουμε μία πτώση στην αλληλευτική δραστηριότητα και όσον αφορά τα διάφορα σκάφη, είτε είναι παραγαδιάρικα είτε όχι, και κυρίως ε, για τα παραγαδιάρικα σκάφη όμως έχουμε σημειώσει πτώση, αλλά ισχύει και για όλα ε, τα υπόλοιπα σκάφη. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουν πέσει ελευτικές δυνατότητες. Do ε, έχει συνέπειες και στην χρηματική αντιπαροχή που δίνεται. Θέλουμε να έχουμε στήριξη του τομέα, η οποία θα πρέπει να είναι πιο αυξημένη. Όσον αφορά τώρα τις αλληλευτικές άδειες, οι αξίες τους ε, επιδεινώνεται αν εξετάσουμε όλα αυτά τα ποσά συγκριτικά, το γεγονός ότι το πρωτόκολλο μόλις εξέπνευσε και το, το γεγονός ότι μας προτείνεται τώρα ένα νέο πρωτόκολλο 6 ετών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές είναι ισορροπημένο. Υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά στις ελευτικές δυνατότητες, ε, τη χρηματική αντιπεροχή, τις ελευτικές άδειες και κάποια πρόσθετα αλλιεύματα. Όλα αυτά ε, δείχνουν ότι προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες, κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχουν ε, λιγότερα λευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει και μια λογική για όλα τα αριθμητικά στοιχεία που μας παρουσιάζονται σε αυτό το πρωτόκολλο. Επειδή λοιπόν υπάρχουν ε, συμφέροντα κατέρωθεν και οι Σεϊχέλες δηλαδή και εμείς ενδιαφερόμαστε και δεδομένου ότι υπάρχει κατάλληλη προσαρμογή όπως σας είπα στις νέες συνθήκες, θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη πρόταση είναι ισορροπημένη. Και επομένως θα είναι χρήσιμη και για τις δύο πλευρές. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Euh, Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας δώσω ορισμένε πρόσθετες πληροφορίες για το πρωτόκολλο αυτό που εγκρίθηκε με την ε, Δημοκρατία των Σεϊχελών πέρυσι. Θα ήθελα να τονίσω τη στρατηγική σημασία που έχει η συμφωνία αυτή και για μας την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλλιευτικούς μας στόλους του τόνου και για τις Σεϊχέλες. Όπως ξέρετε είναι στρατηγική σημασία γιατί πρόκειται για συμφωνία που αφορά αποκλειστική οικονομική ζώνη τεράστια με πολύ μεγάλα αλλιεύματα και επομένως και ό,τι παίζεται χρηματικά εδώ είναι πολύ σημαντικό. Το λιμάνι της Βικτόριας είναι το πρώτο λιμάνι όπου μπορεί να προσεγγίσουν ευρωπαϊκοί στόλοι στον Ινδικό ωκεανό και είναι πολύ σημαντικό για τη διαχείριση των αλλιευμάτων τόνου εκεί. Για την τοπική βιομηχανία επίσης, <clears throat> εκεί υπάρχουν δραστηριότητες ξεφορτώματος και μεταποίησης που γίνονται από τους δικούς μας τόλους και συμβάλλουν και αυτές οι δραστηριότητες στην οικονομική ανάπτυξη τοπικά. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 3.000 θέσεις απασχόλησης υπάρχουν εκεί και τροφοδοτούνται για τη μεταποίηση. Άρα είναι σημαντικό και για μας και για την οικονομία των Σεϊχελών. Για τη δημοκρατία αυτή είναι σημαντική η αναγνώριση του ηγετικού αλλιευτικού ρόλου της Ένωσης εκεί και έτσι ενδυναμώνονται και οι δεσμοί μεταξύ μας. Τώρα τα χαρακτηριστικά του νέου πρωτοκόλλου που εγκρίθηκε όπως είπα τον περασμένο Μάιο έχει ισχύ εξαετή. Και αυτό είναι καλό γιατί ορισμένα άλλα πρωτόκολλα είχαν πολύ χαμηλότερη διάρκεια και έτσι μπορούμε να έχουμε κάποια μεγαλύτερη νομική σαφήνεια, σταθερότητα, ασφάλεια για τη λειτουργία του στόλους μας. Αυτό θέλουν εξάλλου και οι εφοπλιστέ. Και για τις Ιχέλες είναι μια ευκαιρία περισσότερη σταθερότητα στις σχέσεις μας με στις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα ήθελα να επιμείνω στο ότι το νέο αυτό πρωτόκολλο λαμβάνει υπόψη τις προσαρμογές, τις εξελίξεις μάλλον που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ στην εξωτερική της διάσταση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα ως προς τα χρηματοδοτικά τμήματα του πρωτοκόλλου γιατί γενικά η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μειωθεί ενώ των εφοπλιστών έχει αυξηθεί. Για πρώτη φορά λοιπόν εφαρμόζουμε ένα από τα βασικά στοιχεία της διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης της Αλίας που ζήτησαν το Συμβούλιο και το Κενοβούλιο κατά τα διάφορα ψηφίσματα τα περσινά. Πιο συγκεκριμένα τώρα, ποιες είναι οι εξελίξεις που σημειώθηκαν η συμμετοχή της βιομηχανίας που ήταν 35 ευρώ τον τόνο, με αυτό το πρωτόκολλο φτάνει από 55 έως 75 ευρώ τον τόνο. Η βιομηχανία λοιπόν εδώ συμβάλλει πολύ περισσότερο από ό,τι πριν και είναι έτοιμη η βιομηχανία αυτή να συμμετάσχει διότι έχει κέρδη, της αποφέρει κέρδη η συμφωνία. Και από την πλευρά της η Ένωση συμμετέχει ανατόνο 65 ευρώ στο παρελθόν τον τόνο ενώ τώρα 55 με 50. Βλέπετε, θα δείτε ότι Υπάρχει και μια προοδευτικότητα εδώ γιατί στα έξι αυτά χρόνια μέχρι το 19 τελικά στοχεύουμε η βιομηχανία να φτάσει 75 ευρώ τον τόνο και πολύ χαμηλότερη η ενωσιακή εισφορά. Έτσι ανταποκρινόμαστε στις διακυμάνσεις που σημειώθηκαν στην αγορά αλλά και στις δυνατότητες των ε, εταίρων μας. Αυτά όλα προέκυψαν από διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους και τη βιομηχανία, τον τομέα. Για το, τη χωρητικότητα αναφοράς 50.000 τόνοι αυτή τη στιγμή. Το ίδιο με πριν δηλαδή χαμηλή μείωση για να, δούμε, για να ανταποκριθούμε στο πραγματικό επίπεδο των αλλιευμάτων και οι αδειοδοτήσεις της αλλίας επίσης έχουν μειωθεί διότι η προηγούμενη συμφωνία δεν είχε πλήρως χρησιμοποιηθεί. Έξι δυνατότητες αλλίας για τα long liners και 40 για το, τα υπόλοιπα ίδια έτσι ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον της αλίας μας. Επίσης, λάβαμε υπόψη τις δυνατότητες αλίευσης ε, του καθεστώτος της Μαγιότ. Δηλαδή πλοία που ήταν υπό σημαία Μαωρέ, τώρα θα περάσουν σε ευρωπαϊκή σημαία. Μιλήσατε και για την πειρατεία κυρία μου, η οποία οποία εξελίσσεται και αυτή θετικά, δηλαδή μειώνεται. Με 40 τράτες νομίζω ότι φτάνουμε στο μέσο όρο του προηγουμένου πρωτοκόλου που ήταν 25 με 30 αδειοδοτήσεις. Λάβαμε υπόψη μας λοιπόν και τις εξελίξεις και τα περιθώρια ελιγμών που απαιτούνται. Τώρα για τη στήριξη του τομέα, την τομεακή στήριξη. Σφαιρικό ποσό είναι 5.350.000 περίπου. Υπάρχει και εδώ λοιπόν μια προοδευτική αύξηση και αυτό το είχε ζητήσει και οι εκπρόσωποι του τομέα. Το μισό από αυτό το ποσό 2.600.000 για τα πρώτα χρόνια και μετά 2.500.000 δίνονται για την τομεακή στήριξη. Και αυτό δείχνει επίσης την πολύ καλή δυνατότητα απορρόφησης που έχει η χώρα αυτή για την ε, τομεακή στήριξη. Τα προγράμματα που εφαρμόζονται στις Ιχέλες αφορούν κυρίως την ανάπτυξη της τοπικής βιομηχανίας και των τοπικών στολίσκων για τη μεταποίηση. Επίσης υπάρχει σημαντική επένδυση υπέρ του δικού μας στόλου αυτή τη φορά, νέες λιμενικές εγκαταστάσεις δηλαδή με καινούργιες αποβάθρες στο λιμάνι της Βικτόριας. Καλός ρυθμός απορρόφησης λοιπόν και γι' αυτό αποφασίσαμε να συνεχίσουμε σε τόσο ψηλό επίπεδο τη χρηματοδότηση. Να αυτά είναι τα βασικά ως προς το νέο αυτό παροτόκολλο με τις Ειχέλες. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στους ομιλητές. Ο κύριος Άντσες Πρεσέδο καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για την παρουσίασή της και την ε, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευχαριστώ και σας και συμφωνώ με τα όσα είπε η εισηγήτρια για τη συμφωνία με τις Ειχέλες. Ε, η συμφωνία με τις Ειχέλες ξεκίνησε από το 1997. Το πρωτόκολλο το οποίο συζητούμε τώρα έχει τις ρίζες της ε, ε, στην ε, Συμφωνία Συνεργασίας του 2006. Εξέπνευσε πριν από μερικές μέρες η προηγούμενη συμφωνία στις 17 και στις 18 ξεκίνησε η προσωρινή εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου. Η συμφωνία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί συμφωνίζει, συμπληρώνει συγγνώμη, το σύνολο των ε, συμφωνιών που έχουμε για να έχουμε παρουσία στον Ινδικό ωκεανό και κυρίως στο λιμάνι της Βικτόριας που είναι πολύ σημαντικός λιμένας διότι είναι κέντρο επιμελητίας και εκεί γίνεται περίπου το 60% των εκφορτώσεων τόνου του Ινδικού ωκεανού. Ε, πριν από την υπογραφή του πρωτοκόλου ε, πέρασε περίπου ένας χρόνος, έγινε και μία ανεξάρτητη αξιολόγηση και είχαμε σε συνέπεια αυτής της αξιολόγησης μία εντολή η οποία οδήγησε στη διαπραγμάτευση για το πρωτόκολλο. Είναι πολύ θετικά τα όσα συμφωνήθηκαν. Πάντα επιμένουμε ότι οι ελευτικές συμφωνίες ε, χρειάζονται αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε τις κατάλληλες προβλέψεις από πλευράς των ε, του κλάδου για να ε, ξέρουμε εάν επαρκεί αυτός ο χρόνος και ε, πολλές φορές είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που προσφέρεται και δημιουργείται μεγάλη αβεβαιότητα για τις επενδύσεις που μπορούν να γίνουν στον ελευτικό τομέα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, αφορά 46 σκάφη από διάφορες ε, χώρες. Ε, ένα σημαντικό τμήμα θα είναι ισπανικά σκάφη. Θα υπάρξει μία μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα σκάφη και όπως εξήγησε εν μέρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει κάποιος λόγος, αλλά δεν είναι ουσιαστική διαφορά από πλευράς ποσών. Η οικονομική αντιπεροχή είναι ισορροπημένη και φυσικά ακολουθούν και τις συστάσεις της Επιτροπής ε, του Τόνου του Ινδικού Ωκεανού. Θα προσαρμοστούν λοιπόν ε, στα όσα προτείνει οι Περιφερειακές Οργανώσεις Αλίας ε, για τα θέματα αυτά. Και επειδή το θέμα της πειρατείας είναι ευαίσθητο, θα πρέπει να φροντίσουμε οι άδειε οι οποίες δίνονται να μην ε, είναι άδειε οι οποίες μπορεί να ε, δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις για τους ε, πλειοκτήτες. Ως και όδης από πλευρά των σοσιαλιστών επικροτώ τη συγκεκριμένη έκθεση και θα ήθελα να την υποστηρίξουμε εδώ στην έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Λεβίν. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την, την εισηγήτρια για την παρουσίαση της. Τώρα, κάποια παράπονα για τη διαδικασία εδώ ε, που χρησιμοποιήθηκε ε, η Επιτροπή Ανάπτυξης δεν πρόλαβε να εκδώσει ε, γνωμοδότηση για το θέμα αυτό ενώ στο παρελθόν είχαμε πει ότι όλες αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να συνοδεύονται από γνωμοδότηση Επιτροπής Ανάπτυξης. Α, αυτό δεν έγινε εδώ, αυτό δεν είναι σωστό. Τώρα, επί της ε, συμφωνίας αυτής καθεαυτής κατά την άποψή μου πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, αυξάνονται τα τέλη των πλεοκτητών, καλό αυτό. Τώρα, θέλω να ρωτήσω κάτι για τις διάφορες κατηγορίες. Αν υπάρχει, υπάρχει ειδική ποσόστος για καρχαρίες εδώ δεν το είδα. Θυμάμαι ότι στη συμφωνία με τη Μαδαγασκάρη είχαμε μια ειδική ποσόστοση για καρχαριοειδή για καρχαρίες. Φαίνεται ότι είναι μεγάλο παραλίευμα τα καρχαρίες, οπότε ίσως θα πρέπει να υπάρχει και εδώ. Τώρα να θέσω ένα άλλο ερώτημα, ε, διάφορα άλλα θέματα, όχι για αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά για μια άλλη συμφωνία που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή με τις Σεϊχέλες και σχετίζεται με πρόσβαση των Σεϊχελών σε τα μαγιά αλλά επειδή Μαγιότ έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέλος πάντων ευρωπαϊκά υδάτα. Ωραία. Οχτώ των οθυρικά λειτουργούν στα ευρωπαϊκά αυτά είδατε με σημαία σύγχελών. Ερώτηση, ποιος είναι ο πλειοκτήτης αυτών των σκαφών ποια εταιρεία γιατί η Κομισιόν ε, νομίζω αναφέρει κάποια πράγματα σχετικά με το ε, πλειοκτήτη ότι χρειάζεται να υπάρχει μια κάποια τοπική εταιρεία ή εν πάση περιπτώσει κάποιος πίκος ε, εδώ υπάρχει και διμερή συμφωνία με τις Σεϊχέλες τι θα κοστίσει η αλία αυτών των σκαφών με ε, σημαία Αιχελών σε ευρωπαϊκά ύδατα τι άλλες δραστηριότητες αναλαμβάνονται εκεί και κάτι τι άλλο ο τόνος που αλλιεύεται στα ύδατα Μαγιώτο από σκάφη με σε χελών εντάσσεται στις ποσοστώσεις του καθεστώτου ΑΚΕ. Στίβενσον, πρόεδρε, δύο λόγια για την πειρατεία. Γιατί εξ όσων γνωρίζω από τότε που άλλαξε, μια και άλλαξε το πρωτόκολλο όπως είπε και η συγγήτρια, από τότε που άλλαξε το πρωτόκολλο λοιπόν η πειρατεία μειώθηκε στην περιοχή. Και εξ όσων ξέρω εγώ δεν υπήρξε καμία επιτυχής απόπειρα πειρατεία στα τελευταία, τους τελευταίους μήνες. <laughs> ήδη ξέρουμε τι γίνεται στον Ινδικό ωκεανό που υπάρχει μια μονάδα, ομάδα δράσης αν θέλετε που πυροβολεί τις εξολέμβειες των σκαφών των ε, πειρατών ε, και φαίνεται ότι λειτουργεί το, το σύστημα πίστηκαν πολλοί ε, που θα είχαν πρόθεση να κάνουν πειρατεία στον Ινδικό ωκεανό να μην το κάνουν. Και η κυβέρνηση της Σομαλίας, γιατί εκεί ήταν χειρότερα τα πράγματα, ήρθε σε επαφή μαζί μου ρωτώντα κατά πόσον είναι δυνατόν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για μια συμφωνία ε, ε ακτίνα 12 ναυτικών μιλίων γιατί θεωρούν ότι ελέγχουν την πειρατεία αυτή τη στιγμή. Εγώ υποστηρίζω την έκθεση πάντως. Κυρία Φράγκα. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Πατράου. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική αυτή η συμφωνία. Έχει γίνει πολύ καλή διαπραγμάτευση και χαίρομαι που έχει διαρκεία 6 ετών, ε, που θα δούμε σε λίγο ότι με τις κομόρες δεν ε, συνέβη, παρά το γεγονός ότι στην έκθεση αξιολόγηση η πρόταση ήταν για 6 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση το καταφέραμε και αυτό σημαίνει ότι ο κοινοτικό ε, στόλος μπορεί να προγραμματιστεί και να προετοιμαστεί καλύτερα για το μέλλον. Εγώ με κάποιους, όπως η κυρία Ρόντουστ, μεταβήκαμε στις Σεϊχέλες με αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας και Χαίρομαι καταρχάς ε, που ε, έχει ολοκληρωθεί ο νέος λιμένας χάρη στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση η τομεακή στήριξη χρησιμοποιήθηκε όπως ε, επιθυμεί ο Θεός, όπως ήθελαν οι Σεϊχέλες και όπως ήθελε και ο κοινοτικό κλάδος διότι όσοι ήμασταν εκεί είδαμε ότι το λιμάνι της Βικτόρια που είναι ο πιο σημαντικός λιμένας στην περιοχή ε, είναι ε, λιμάνι στο οποίο αποτελεί απόλυτη συμφόρηση και το γεγονός ότι θα έπρεπε να συγχρονιστεί αυτός ο λιμένας είναι κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό και για τις δύο πλευρές. Δεύτερον, χαίρομαι διότι ε, όταν πήγαμε εκεί μας είπαν οι ναυτικοί τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ε, κόσμος ο οποίος ε, να ασχολείται με την αλληλεία διότι το μεγαλύτερο τμήμα του εργατικού δυναμικού είναι ε, ε, στον τομέα του τουρισμού. Επομένως, η μόνη λύση είναι να χρησιμοποιούν ένα ελάχιστο τμήμα ανθρώπων που είναι διατεθειμένοι ε, να εργαστούν στα σκάφη αυτά και πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι ελάχιστα καταρτισμένοι, ανειδίκευτοι σχεδόν και ας είπαν οι πλειοκτήτες ότι είναι δύσκολο να προσλάβουν αυτούς τους ανθρώπους στα σκάφη τους διότι ε, συνήθως, ε, λοιπόν, επειδή δεν βρίσκουν, έχουν ε, ναυτικούς από χώρες ακές, κυρίως ενεγαλέζους, που είναι άρθροι, ακαταρτισμένοι και ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά και έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα να προσλάβουν ανειδίκευτους ε, από τις Σεϊχέλες. Στη συμφωνία έχει γίνει λοιπόν κάτι πάρα πολύ καλό. Καταρτίζεται ένας κατάλογος στον οποίο καθορίζεται τι κατάρτιση θα πρέπει να έχουν οι ναυτικοί και σε περίπτωση που οι εφαπλιστέ ε, απαιτούν ε, ε, κάποια μορφή κατάρτιση που δεν περιλαμβάνεται σε αυτό τον κατάλογο, αποκλείονται από τη χρηματοδότηση και αυτό είναι θετικό γιατί στο παρελθόν δεν είχε κανένα νόημα αυτό το οποίο προβλεπόταν. Υπάρχει και το θέμα της Μαγιώτ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το πρόβλημα με τη νομική βάση ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απαράδεκτη, διότι ε, γίνεται διαπραγμάτευση για μια ελευτική συμφωνία ε, που κάνει το Συμβούλιο και μάλιστα υπήρχε και μια αντίστοιχη περίπτωση στο παρελθόν ε, η οποία εκδικάστηκε στο δικαστήριο. Η νομική βάση δεν είναι σωστή. το είπε και η κυρία Πατραωνεύος. Υπάρχουν λοιπόν οι ερωτήσεις μου. Ελπίζω να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Οι πλειοκτήτες είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με αυτή τη συμφωνία. Και ε, μου άρεσε και αυτό που είπε ο κύριος Στίβενσον για τη Σομαλία, διότι αν θυμάστε καλά πάντα μας κατηγορούσαν εμά που ασχολούμαστε με την αλία ότι η πειρατεία προέκυψε γιατί γινόταν υπερεκμετάλλευση από πλευράς ε, κοινοτικού στόλου ε, για τις αλληλευτικέ δυνατότητες τη Σομαλία. κάτι το οποίο ήταν απόλυτα ψευδέ. Χαίρομαι λοιπόν που ζητούν τώρα συμφωνία για να αντιμετωπίσουν την πειρατεία. Δείχνει πόσο μεγάλες αντιφάσει πολλές φορές πρέπει να ζήσουμε εμεί στον κόσμο της, πειρα... της αλληλείας. Πολλές φορές είναι παράλογα όλα αυτά τα πράγματα. Κύριε Ρόντους. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα συμπληρωματικά να πω ότι πολύ συχνά επικρινόμεθα ότι κάνουμε ταξιδάκια ε, και εκδρομές. Ε, πήγαμε στις Σεϊχέλες ε, αλλά για συγκεκριμένο σκοπό. Θα θυμάστε ότι παλιότερα είχαμε συζητήσει με τον τόνο ο, είχαμε ε, πει ότι για τα τονοθυρικά ήταν κρίμα που δεν υπήρχαν φωτοβολταϊκά στη σκεπή των σκαφών ε, και μια μικρή εταιρεία της περιοχής μου ε, ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα στις Αιχέλες και έφτιαξε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πάγωμα, για την κατάψυξη του τόνου ε, το ανέπτυξαν το σύστημα αυτό και χρησιμοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία ε, και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Ρόντουστ. Ε, δεν έχει δει κάποιο άλλο το λόγο. Να δώσω λοιπόν καταρχάς το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στις ερωτήσεις και μετά στην εισηγήτρια για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Θα προσπαθήσω πάντως να απαντήσω στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Πρώτα-πρώτα για τους καρχαρίες. Δεν ε, ε αλλιεύονται καρχαρίες στην περιοχή ε, και δεν αναφέρονται γι' αυτό καθόλου στις ε, στη συμφωνία, στο πρωτόκολλο γιατί τα παραγαδιάρικα δεν ε, ε, περιλαμβάνονται ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν μεγάλο ρόλο να παίξουν ε, όσον αφορά τις ε, οπότε η αλία εχουν μεγάλη ρολο να παιξουν οσον αφορα τελείως τυχαία και πολύ μικρή σε ποσότητα Τώρα, για μια, θα πω δύο λόγια για μια άλλη εταιρή, ε, συμφωνία που αναφέρθηκε προηγούμενα που σχετίζεται με την πρόσβαση των σκαφών με σημαία σε χελών στα τα Μαγιότ. Έγινε αυτή η συμφωνία γιατί διότι θεωρήσαμε ότι ήταν η νομική υποχρέωσή μας η αρμοδιότητά μας για τα ύδατα αυτά ε, συνεπάγεται και την υποχρέωση να συναυθεί μια τέτοια συμφωνία. Οι όροι τώρα της συμφωνίας αυτής είναι παρόμοιοι με παλιότερες συμφωνίες ε, ιδιωτικής φύσεως ε, χρηματική αποζημίωση αλλά από τους εμπόρους έτσι δεν είναι από την... είναι τελείως εμπορική συμφωνία η οποία δεν ε, ε, είναι ιδιωτικού δικαίου Θα συζητήσετε μελλοντικά φαντάζομαι για την ε, συμφωνία αυτή οπότε μπορούμε να τη ε, συζητήσουμε περαιτέρω και πιο λεπτομεριακά τη συμφωνία αυτή. Θα μπορώ να τα συζητήσω αυτά διμερώς και με την κυρία Λεβίν. Τώρα ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια ε, που μας δώσατε για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κομισιών και Σύχελων. Ευχαριστώ. Η κυρία Πατρά τώρα. Alguns comentários relativamente aos, eh, às observações feitas. Eh, Δεν έχω ε, πολλά να προσθέσω σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Όμως ε, έγιναν κάποιες θα ήθελα να αναφερθώ στον αριθμό των σκαφών ο οποίος μειώθηκε γιατί διότι οι άδειε που είχαν δοθεί με το προηγούμενο πρωτόκολλο δεν εξαντλήθηκαν και μία από τις αναπροσαρμογές που έγινε ήταν η μείωση του αριθμού των σκαφών. Τώρα αυτά που είπε ο κύριος Στίβενσον γιατί για την ε, πειρατεία ότι μειώθηκε η δραστηριότητα αυτή αυτό είναι αλήθεια παρόλα αυτά θεωρούμε ότι γίνονται απόπειρες πειρατείας πολλές στην περιοχή χτες έμαθα ότι στην ακτή της Λουάντα εξαφανίστηκε λιβεριανό σκάφος πράγμα που σημαίνει ότι συνεχίζουν να είναι ενεργοί οι πειρατές στην περιοχή στις Αιχέλες μπορεί να έχουν χημειωθεί η δραστηριότητα αλλά στην περιοχή όχι είναι γεγονός ότι ε, λαμβάνονται μέτρα για το ε, κατά της πειρατείας αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για σημαντικές επιτυχίες εκεί. Η Ζαμπέλα μίλησε για τη διαδικασία και είπε ότι η Επιτροπή ΔΕΒΕ δεν έχει νομοδοτήσει. Ωραία, το, εντάξει αλλά δεν νομίζω ότι φταίμε εμείς επειδή δεν γνωμοδότησε η Επιτροπή Ανάπτυξης άμα η Επιτροπή δεν θέλει να γνωμοδοτήσει δεν προλαβαίνει να γνωμοδοτήσει τι να κάνουμε θα μπορούσε να έχει γνωμοδοτήσει κατά την άποψη μου η Επιτροπή Ανάπτυξης δεν ήθελε να το κάνει δεν νομίζω ότι παρεμποδίζουμε κανέναν να εκφραστεί Όποιος θέλει να ακουστεί φωνάζει. Αναφέρθηκαν και άλλα θέματα δεν αναφέρθηκαν τώρα οι καρχαρίες τι γίνεται με τους καρχαρίες δεν περιλαμβάνεται τίποτε εδώ υπάρχουν ε, βεβαίως υπάρχουν 300 είδη καρχαριών αλλά εδώ δεν φαίνεται να γίνεται μεγάλη αλίευση κανενός είδους ε, καρχαριών. Τώρα αν θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για τις επιπτώσεις στη βιωσιμότητα θα πρέπει να γίνουν επιστημονικές μελέτες στην περιοχή. Τώρα για την κρόαση για την ε, για αυτά που είπε η Κομισιόν θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν αναφέρθηκα σε νούμερα στην παρουσίασή μου γιατί πραγματικά η, αλλη... η αλληλεία μπορεί να είναι σημαντικός κλάδος για τις Αιχέλες αλλά δεν είναι ο πλέον σημαντικός από οικονομική άποψη. Σκέφτηκα λοιπόν να μην παρουσιάσω σχετικούς αριθμούς γιατί ξέρω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις για τα νούμερα. Προσπάθησα να αναφέρω ποιοτικά στοιχεία και όχι τόσο ποσοτικά στοιχεία της συμφωνίας. Ευχαριστώ πάντως για τις παρατηρήσεις που κάνατε και ελπίζω να γίνουν και άλλες ε, να περάσει η έκθεση αυτή ε, χωρίς άλλα σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πατρά. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Διεθνή Σύμβαση του Διεθνού ε, Ναυτιλιακού Οργανισμού του 1995 για τα πρότυπα εκπαίδευση, έκδοση πιστοποιητικών και τήρηση φυλακών για το προσωπικό των ελευτικών σκαφών. Ε, έγινε μια παρουσίαση, έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και τώρα η συντάκτρια της γνωμοδότησης, η κυρία Ζαμπελτομά, θα μας κάνει την ε, παρουσίαση της γνωμοδότησής της. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει λοιπόν να εγκρίνει, να επικυρώσει την διεθνή αυτή σύμβαση που θα γίνει τελικά το ελάχιστο διεθνές πρότυπο για την πληροφόρηση των αλλιέων και για όλους τους εργαζόμενους στα αλλιευτικά πλοιάρια. Η σύμβαση αυτή συμπληρώνει την προηγούμενη για την εμπορική ναυπητηλία που είχε εγκριθεί από την STSWF στο Λονδίνο με 74, από 74 κράτη μεταξύ των οποίων και τα περισσότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βασική, το βασικό κριτήριο που προτείνει είναι να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων και για τα πρόσωπα και για τα αγαθά αλλά και για το περιβάλλον. Η αλληλευτική δραστηριότητα όπως ξέρετε είναι η πιο επικίνδυνη οικονομική δραστηριότητα από όλες. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη θνησιμότητα. Θα σας δώσω δύο ρυθμούς. Το 11 στη Γαλλία 32 πλοιάρια ε, υπέστησαν βαριά ατυχήματα, στην Ισπανία 38. Κάθε χρόνο σημειώνονται θάνατοι σε μεγάλο αριθμό. Υπάρχουν λοιπόν νεκροί αλλά και άλλα εργατικά ατυχήματα, εργασιακά ατυχήματα, πολύ σοβαρά όπως ε, ακροτηριασμοί κλπ. Η επικύρωση λοιπόν από τα κράτη-μέλη της σύμβασης αυτής πρέπει να εγκριθεί και από την Ένωση, να επικυρωθεί, και περιέχει μια ειδική ρήτρα που λέει ότι σε περίπτωση διαφορών μεταξύ χωρών μελών υπερισχύει η ενωσιακή νομοθεσία. Τα κράτη-μέλη που έχουν ήδη επικυρώσει πρέπει να υποβάλουν στο Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης σημείωμα που να αναφέρει ότι περισχύει το ενωσιακό δίκαιο. Φυσικά πρόκειται για κάποιο, κάποιο πρόοδο διεθνώς διότι μάλλον θα βελτιώσει τους όρους ασφαλείας, ασφαλούς εργασίας στα αλληλευτικά πλοία και θα μειωθούν τα ατυχήματα. Δεύτερον, θα εναρμονίσει προς τα πάνω τα απαιτούμενα επίπεδα κατάρτισης Παρόλα αυτά υπάρχουν και μερικές ελλείψεις. Πρώτον, η σύμβαση δεν αφορά παρά μόνον τα πλοιάρια άνω των 24 μέτρων και τα υπόλοιπα δεν λέει τίποτα. Τίποτα δεν προβλέπεται για τα μικρότερα. Ενώ γνωρίζουμε ότι τα μικρότερα αυτά πλοιάρια είναι τα περισσότερα και επίσης τα σημαντικότερα όλου, σε όλο τον ευρωπαϊκό στολίσκο. Άρα τελικά η σύμβαση αφορά πολύ λίγους από τους συνολικά εργαζόμενους στην Αλία. Δεύτερον, υπάρχουν ελλείψεις ακόμη και για αυτά που προβλέπονται για τα μεγάλα πλοιάρια. Έπειτα, Επιταλέγω, αν και δεν ήταν αυτός ο στόχος, θα έπρεπε να πούμε ότι δεν μιλάει καθόλου για τις συνθήκες εργασίας και ασφαλείας πάνω στα πλοία. Ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι οι συνθήκες εργασίας και ασφαλείας, ιδίως τη νύχτα, είναι πολύ σημαντικό θέμα Γι' αυτό εξάλλου υπενθυμίζουμε ότι η Σύμβαση 188 πρέπει και εκείνη να συμπεριληφθεί στην κοινοτική νομοθεσία. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η ποιότητα και ο βαθμός εξυγχρονισμού των πλοιαρίων παίζουν και αυτά κάποιο ρόλο στην ασφάλεια και ότι δεν υπάρχουν σχετικώς πρότυπα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς το λόγο. Κανείς, ε, ούτε κομισιόν, από ό,τι βλέπω. Παρακαλώ. Ε, ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω την συντάκτρια της γνωμοδότησης για την γνωμοδότησή της, για το γεγονός ότι υποστηρίζει την πρότασή μας, όπως επεσήμανε και πάλι. Ο τομέας της είναι είναι τομέας ε, στον οποίο έχουμε αρκετά ατυχήματα και αν δείτε τι γίνεται στην έκθεση, τα περισσότερα ατυχήματα είναι ε, ανθρώπινο σφάλμα. Επομένως η κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει ερώτηση της εισηγήτριας γιατί περιορίζουμε ε, το κείμενο απλώ ε, στην κύρωση της σύμβασης και δεν έχουμε ένα κοινοτικό κείμενο όπως έχουμε κάνει σε άλλες περιπτώσεις. Στην αρχή είχαμε, προτείνει, ε, είχαμε σκεφτεί το ενδεχόμενο να προτείνουμε οδηγία όπως έχουμε κάνει σε άλλες περιπτώσεις αλλά τελικώς καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν αξίζει τον κόπο γιατί είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ναυτικών που ε, τους αφορά αυτή η σύμβαση και τα όσα ισχύουν στη χώρα μας ούτως ή άλλως ε, ως πρότυπα ασφαλείας είναι πολύ πιο αυξημένα από αυτά που έχουμε στις διεθνείς συμβάσεις. Ε, η σύμβαση εφαρμόζεται για τα σκάφη των 24 μέτρων και άνω. Ε, κάτω από τα 24 μέτρα ισχύει η εθνική νομοθεσία και οι συνθήκες τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο αυξημένα τι ε, γίνεται τώρα όσον αφορά την κύρωση. Εμείς ε, θεωρούμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κυρώσουν τη σύμβαση, όπως ε, τους ενθαρρύνουμε άλλωστε να κάνουμε, και εφαρμόζοντας όσον αφορά την εσωτερική κινητικότητα την Οδηγία 2036, δεν θα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα. Ε, μία ακόμα σημαντική παρατήρηση της εισηγήτριας είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ της έκθεσης αυτής και της έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την Αλία. Αυτές είναι οι δύο πιο σημαντικές ε, συμβάσεις για τον ε, τομέα της Αλίας και συμπληρώνουν η μία την άλλη. Όσον αφορά την... 188 τη Σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο άρθρο της συνθήκης, το άρθρο 55, το οποίο επιτρέπει τη σύμβαση, όπως γίνεται και με τους ναυτικούς ε, που έχει δοθεί η δυνατότητα να εγκριθεί ε, και υπάρχει συμφωνία μεταξύ ε, κοινωνικών εταίρων. Όσον αφορά τώρα τη στήριξη που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα λευτικά σκάφη, να σας υπενθυμίσω ότι το Ταμείο Αλληλείας ε, που ισχύει τώρα αλλά και το μελλοντικό Ταμείο Αλληλείας προβλέπει στήριξη για τον εξυγχρονισμό και ε, την ασφάλεια και την υγιεινή επί του σκάφους, όπως επίσης και την επαγγελματική κατάρτιση. Επομένως, ε, μπορεί να δοθεί η χρηματοδότηση για καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση και προβλέπεται αυτό από τα ταμεία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητά τον λόγο. Κυρία Τόμα, θέλετε να κάνετε κάποια άλλη παρατήρηση. Όχι, ωραία, να περάσουμε στο επόμενο. Ευχαριστώ, όλα καλά. Τίποτα, τίποτα. Θα Ήθελα να πω ότι είμαι ευχαριστημένη. Εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Σημείο 16, Πρωτόκολλο Ευρωπαϊκής Ένωσης Κομορών σχετικά με τον καθορισμό των ελευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπεροχής που προβλέπονται στη Συμφωνία... Α, συγγνώμη. Προθεσμία για τις κατάθεση τροπολογιών 27 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι. 27 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι, τροπολογίες για το προηγούμενο θέμα. Στο 16 λοιπόν, θα έχουμε την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, πρόταση και ως συνήθως ε, στη συνέχεια θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή, τον κύριο Βαλέσα. Να δώσουμε λοιπόν πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας εξηγήσει λίγο τις διαπραγματεύσεις και την πρόταση και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή και στους υπόλοιπους βουλευτές. Κομισιόν. Merci beaucoup, <clears throat> Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για τις Κομόρες λοιπόν. Υπάρχει επίσης ένα νέο πρωτόκολλο που το διαπραγματευτήκαμε πέρυσι. Επικυρώθηκε στις 5 Ιουλίου. Πρόκειται βέβαια για συμφωνία που δεν έχει μεγάλη σχέση με εκείνο των για με εκείνη των Σεϊχελών. Δεν είναι η ίδια η σημασία της, υπάρχει πολύ μικρότερος στόλος. Αλλά παρόλα αυτά συμπληρώνει το σύνολο του, των συμφωνιών που έχουμε συνάψει στον Ινδικό ωκεανό. <clears throat> Είναι λοιπόν σημαντικό για να διασφαλίσουμε και την συνέχεια της πολιτικής αυτής στον Ινδικό ωκεανό. Το διαπραγματευθήκαμε, διαπραγματευόμασταν επί τρία χρόνια. Θέλαμε μεγαλύτερη διάρκεια από τα προηγούμενα, όπως και για τις Ειχέλες. Αλλά παρά όλες μας τις προσπάθειες, οι Κομόρες δεν δέχτηκαν δέσμευση πέρα από τα τρία έτη. Κρίμα γιατί με μεγαλύτερη διάρκεια θα είχαμε προχωρήσει περισσότερο και στη συμβολή μας, στη χρηματική. Τέλος πάντων, αυτό βγήκε από τη διαπραγμάτευση. Τώρα τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας αυτής όπως και με τις Ειχέλες εφαρμόσαμε τις αρχές της ε, μεταρρύθμισης της ΚΑΛΠ και άρα οι εφοπλιστές από 35 αύξησαν τη συμβολή τους πολύ και οι καταποκοπήν πληρωμές επίσης έφτασαν το 12% η συμβολή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μειώθηκε από 65 ευρώ τον τόνο σε 50. Άρα και σε αυτή τη διαπραγμάτευση μπορέσαμε να εφαρμόσουμε αυτές τις βασικές αρχές της μεταρρύθμισης. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία της βέβαια, όπως η ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και με τις Σεϊχέλες. Τώρα εφαρμόζεται παντού, σε όλα τα πρωτόκολλα. Επίσης, είναι λίγο πιο τεχνική η συμφωνία γιατί εφαρμόζεται τώρα προοδευτικά το σύστημα ηλεκτρονικής αναφοράς, το λεγόμενο ERS που επιτρέπει πολύ πιο αξιόπιστο και ακριβή έλεγχο των παλιευμάτων είναι σύστημα που εφαρμόζεται ήδη στους ευρωπαϊκούς στόλους και πιέζουμε τους εταίρους μας να το εφαρμόσουν και αυτή ένα ηλεκτρονικό δηλαδή σύστημα. Θα γίνει αυτό σε μερικά χρόνια, ανάλογα με τις δυνατότητες των κομμωρών. Θα γίνει όμως. Και έτσι θα μπορούμε να παρακολουθούμε πολύ πιο αξιόπιστα τα αλλιεύματα άλλα χαρακτηριστικά. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα η χωρητικότητα είναι 6.000 τόνοι και εδώ λάβουμε υπόψη μας τις εξελίξεις στον Ινδικό ωκεανό δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα αλλιευτικά πλοιάρια από πριν και εδώ συγκρίναμε με την κατάσταση στη Μαγιότ και τις εξελίξεις ως προς την πειρατεία. Ο αριθμός των αδειών είναι σταθερός από 45 σε 42 για τις τράτες. 45 ήταν λίγο υπερβολικός αριθμός και για τα υπόλοιπα μειώσαμε από 25 σε 20. Αλλά και αυτό αρκεί. Μεγαλύτερη αριθμία από τις Σεϊχέλες γιατί υπάρχει εκεί ο γαλλικός στόλος στη Ρεουνιόν. En partie, euh, en grande partie même je dirais, Για τα παραγαδιάρικα που αλλιεύουν ξυφίες. Και πήραμε υπόψη μας και το θέμα των καριχαριών. Τέλος για το συνολικό ύψος της εισφοράς μας 600.000 ευρώ το χρόνο και τα μισά από αυτό το ποσό είναι για την τομεακή στήριξη. Δεν είναι πολύ ψηλά ποσά γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη τέτοιας χρηματοδότησης και έχουν και πολύ λίγες διοικητικές δυνατότητες και το λάβαμε και αυτό υπόψη μας. Αυτά κυρίες και κύριοι βουλευτέ είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου αυτού πρωτοκόλλου με τις Κομόρες. Ευχαριστώ κύριε Βαλέσα. Dziękuję panie przewodniczący. Ten protokół zapewnia możliwości połowowe dla floty. Ευχαριστώ πολύ. Το πρωτόκολλο αυτό εγγυάται ε, δυνατότητες αλίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτε το παράξενο νομίζω ότι θα πρέπει να το εγκρίνουμε η παρουσίαση που έγινε ε, από την Κομισιόν ήταν ε, αρκετά εκτενής ε, εκτενής και ε, γι' αυτό δεν έχω τίποτα να συμπληρώσω. Σας λέω απλώς ότι η ποσότητα που καλύπτεται σημαίνει ότι γύρω στα 42 σκάφη θα μπορούσαν να αλλιεύουν στην περιοχή. Από το 2000 παλιότερα ήταν πολλά τα σκάφη που ήταν στην περιοχή από το 2005 και δόθε λόγω της πειρατείας ε, στην περιοχή ο αριθμός των σκαφών μειώθηκε ε, και γι' αυτό και εμείς ε, πιστεύουμε ότι το πρωτόκολλο αυτό καλύπτει επαρκή αριθμό σκαφών, δίνει θέσεις εργασίας. Σας ζητώ να το υποστηρίξετε. Η κυρία Φράγα. Ε, ναι, ευχαριστώ. Δύο θέματα. Το ένα το ανέφερα ήδη, το θέμα των εξετών είναι σημαντικό γιατί η έκθεση ε, του εκ των υστέρων ή εκ των προτέρων ε, ελέγχου, δεν ξέρω πώς να τον αποκαλέσω, είναι πολύ σημαντική και φαίνεται ότι υπήρχε συμφωνία να είναι έξι χρόνια. Φαίνεται τελικά δεν τα καταφέραμε. Οι κομόρες για κάποιο λόγο δεν θέλουν να συνάψουν συμφωνία 6 ετών. Και μετά υπάρχει το θέμα των ναυτικών πρέπει, ε, λέγεται, να έχουμε ναυτικούς από τις Κομόρες. Δεδομένης όμως της κατάστασης ε, στις Κομόρες, είναι πολύ μικρή αλληλευτική διαστηριότητα. Δεν υπάρχουν λιμένες τους οποίους μπορούν να ε, μπαρκάρουν και να ξεμπορκάρουν οι ναυτικοί. Ε, νομίζω ότι ο, ο κανονισμός στη συμφωνία αυτά τα οποία προβλέπει δεν είναι σωστά. Θα έπρεπε όπως είχαμε κάνει ε, και στις προηγούμενες συμφωνίες να έχουμε και τη δυνατότητα να έχουμε ναυτικούς ε, χωρών ΑΚΕ και έτσι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την, τη συγκεκριμένη περίπτωση των ε, ναυτικών από τις Κομόρες. Και θα ήθελα να μου εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπάρχουν αυτοί οι όροι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν. Είναι πολύ μικρό ε, το χρονικό διάστημα και δεν υπάρχουν κατάλληλες λιμενικές δομές για να μπορέσει κάποιος ε, να εκφορτώνει καταλήλως. Στην προηγούμενη συμφωνία που είδαμε για τις Σεϊχέλες, ε, μπορέσαμε να έχουμε ένα προσανατολισμό για το μέλλον και ένα περιφερειακό προσανατολισμό και νομίζω ότι αυτό είναι ο σωστός προσανατολισμός για τους ε, ε, παρατηρητές που θα θέλαμε να έχουμε στο μέλλον. Ε, δεν μου αρέσει η συμφωνία για τους ναυτικούς, γιατί δεν έχουμε μια συμφωνία και, και θέλω να ξέρω και τι έγινε στο τέλος με αυτά τα έξι χρόνια, γιατί δεν μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί έξι χρόνια. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ε, κάποια άλλη παρέμβαση, κυρία Λεβίν. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Βαλέσσα για την παρουσίαση. Συγκεκριμένο ερώτημα σχετικά με τη ρήτρα αποκλειστικότητα. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια ρήτρα και σε αυτήν εδώ τη συμφωνία Ξέρω ότι υπάρχει μια συμφωνία ε, μεταξύ Ισπανίας και Κομορών σχετικά με πέντε αλλιευτικά σκάφη και γι' αυτό το λέω θα πρέπει να υπάρχει μια ε, η συμφωνία με την Ισπανία είναι ιδιωτική έτσι ε, και εκεί τα σκάφη αλλιεύουν σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους και τα λοιπά. Η Κομισιόν το ξέρει αυτό μπορεί να μας πει αν ενημερώθηκε από το κράτος μέλος την Ισπανία Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν ή θα ήθελα, ε, τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να ενημερώνουν την Κομισιόν. Η Κομισιόν θα επρεπε να βάλει ένα σχετικό όρο σε κάποιους κανονισμούς, δεν τα κατάφερε, δεν ξέρω. Ε, λοιπόν, τι ξέρει σχετικά η Κομισιόν ε, ή για αυτή την υπόθεση με την Ισπανία ή με, για άλλες συμβάσεις, συμφωνίες με τις Κομόρες στον Ινδικό ωκεανό. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν να απαντήσει. Oui, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Πρώτα πρώτα για τον αριθμό των σκαφών που προβλέπονται. Είναι γεγονός ότι παλιά είχαμε 40 και 25 ε, περάσαμε στα 42 και 20 μειώθηκε ο αριθμός των σκαφών αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα διαπιστώσαμε ότι ε, λιγότερα σκάφη χρησιμοποιούσαν τη συμφωνία από ό,τι στο παρελθόν γι' αυτό ε, μειώσαμε τον αριθμό των αλλιευτικών σκαφών στην καινούρια συμφωνία αλλά αυτό επαρκεί ή δεν πρόκειται να υπάρχουν περισσότερα σκάφη που θέλουν να πάνε και να αλλιεύσουν μην ανησυχείτε και θα πρέπει να υπάρχει και μια συνέχεια με τις διάφορες, στις διάφορες συμφωνίες βεβαίως Τώρα, από εκεί και πέρα και στην έκθεση αξιολόγησης και εμείς και τώρα ελέγξτε ότι θα θέλαμε αν ήταν δυνατόν διάρκεια συμφωνίας μεγαλύτερη, 4, 5, 6 χρόνια. Πάνω από 3 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά στις διαβουλεύσεις, στις διαπραγματεύσεις, δεν ήταν τόσο εύκολο όπως ελπίζουμε. Και ε, για τις Κομόρες ήταν αδιανόητο να υπογράψουν πρωτόκολλο πέρα από τρεις, ε, ε, τρία έτη. Ε, προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ότι αυτά σήμαινε περισσότερα χρήματα ε, ε, για τον στόλο και τα λοιπά, θα βοηθούσε οικονομικά ή δεν το καταλάβαιναν δεν ξέρω αν ήταν πολιτικές οι, οι αιτίε πάντως ήταν πάρα πολύ έντονη η αντίδρασή τους επέμεναν ότι δεν θέλουν να διαπραγματευτούν για πάνω από τρία χρόνια για, αν επιμέναμε στα έξι χρόνια θα μπλοκαριζόταν η διαπραγματεύση τώρα για τους ναυτικούς ε, τους αλείς δεν ξέρω δεν είναι. Είχα λάβει μέρος στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις αλλά για παραδοσιακούς λόγους γινόταν αυτό και στις παλιότερες συμφωνίες υπήρχε ο όρος να απασχολούνται ε, κομοριανοί Επιέμενε λοιπόν να ανα Επέμεινε λοιπόν η άλλη πλευρά να διατηρηθεί ο όρος αυτός και υπαναχωρήσαμε αν θέλετε, το δεχτήκαμε κι εμείς. Τώρα, όσον, άμα δούμε τις λεπτομέρειες, ε, τρομερό, γιατί οι ναυτικοί αυτοί από τις κομμόρες πρέπει να απασχοληθούν, είναι ένας όλος και όλος και υπάρχει όλα η δυνατότητα οι πλειοκτήτες να ε, καταβάλουν ένα ποσό λογικό ε, ως τιμωρία αν θέλετε τρόπον την λοιπόν μην ανησυχούμε ιδιαίτερα γι' αυτό το αυτόν τον όρο αλλά σε γενικές γραμμές ο, θα προσπαθήσουμε μάλλον προσπαθούμε μέσα του πρωτοκόλλου να προωθήσουμε την απασχόληση ναυτικών από τις χώρες ΑΚΕ η κυρία Φράγκα για τους παρατηρητές που αναφέρθηκα. Είναι γεγονός. σωθούμε να οργανώσουμε τα σχετικά και θέλουμε αν είναι δυνατόν περιφερειακούς παρατηρητές σε περιφερειακό επίπεδο ε, προσπαθούμε, αυτό το προσπαθούμε να προωθήσουμε ούτω ώστε να μην υποχρεωμένα τα σκάφη να πάνε στο λιμάνι για να μπαρκάρει κάποιος παρατηρητής και μετά να πάνε να τον, ε, για να ξεμπαρκάρει κτλ. κτλ. Επιμείναμε λοιπόν στις συζητήσεις μας στο γεγονός ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παρατηρητές περιφερειακή. Τώρα, για τη ρήτρα αποκλειστικότητα που είπε η κυρία Λεβίν, μα είπε ότι δεν υπάρχει στο πρωτόκολλο. Λάθο, κυρία μου, ίσω δεν ψάξατε αρκετά. Στο πρώτο άρθρο Στη τρίτη παράγραφο αναφέρονται ακριβώς τα της αποκλειστικότητας. Επίσης και στην συμφωνία αναφέρονται σχετικά. Μπορεί να μου πείτε ότι είναι πειραιητό να αναφέρονται δύο φορές, ωστόσο αναφέρονται. Δεν πειράζει που ναι, αναφέρονται δύο φορές. Είναι λοιπόν υφίσταται η ρήτρα αποκλειστικότητα σαφέστατα και αυτό καλύπτει και τις περιπτώσεις των ιδιωτικών αδειών και λοιπά που αναφέρεται. Δεν γνωρίζω την ε, ε, συγκεκριμένη προς ε, συμφωνία που αναφέρατε για ένα κράτος μέλος με εκπλήσει αυτό που λέτε αλλά ρήτρα αποκλειστικότητας υπάρχει. Είδου οι απαντήσεις που έχω να δώσω και σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που θέσατε. Ευχαριστώ κυρία Φράγα. Εγώ για να καθησυχάσω την κυρία Λεβίν, να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένα ισπανικό ή γαλλικό σκάφος ή από οποιαδήποτε εθνικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει ιδιωτικές συμφωνίες με τις Κομόρες. Πρόκειται για σκάφη των Σεϊχελών. Αυτά είναι τα σκάφη που έχουν συμφωνίες με τις Κομόρες, αλλά είναι ε, σκάφη με σημαία Σεϊχελών. Αυτό πρέπει να είναι σαφές και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε εξηγήσει ε, πάρα πολλές φορές και για τα αθηνοειδή και για τα αθηναλιευτικά. Δεν είναι σκάφη τα οποία έχουν σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σκάφη τα οποία έχουν σημαία Σεϊχελών και δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένει η κυρία Λεβίν. Κάποιος άλλος, ο κύριος Βαλέσα, α, συγγνώμη, κυρία Λεβίν. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω την κυρία Φράγα για τη διευκρίνηση. η διοργάνωση δηλαδή των μεγάλων ε, ε ψυγείων θυναλιευτικών αλλιεύει με σε ηχελών. Αυτό είναι σαφές. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για αυτές τις ιδιωτικές συμφωνίες, γιατί εμείς προσπαθούμε να το συμπεριλάβουμε αυτό στην εξωτερική ε, διάσταση της κοινή ελευτικής πολιτικής και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, βρίσκει σύμφωνο και το Συμβούλιο. Έχει ήδη συμφωνήσει το Συμβούλιο σε αυτό. Ναι, η Κομισιόν. Όπως σας είπε και η κυρία Φράγκα, δεν πρόκειται για σκάφη με σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα οποία αλλιεύουν με αυτές τις ιδιωτικές συμφωνίες. Δεν αφορά άμεσα λοιπόν την εφαρμογή του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν σκάφη από διάφορες χώρες που αλλιεύουν στα ύδατα των Κομορών. Ε, κάναμε μια αξιολόγηση, έχουμε μια εικόνα για τα διάφορα σκάφη. Υπάρχουν ασιατικά, αφρικανικά σκάφη, σκάφη με διάφορες σημαίες που αλλιεύουν στην ε, ε, περιοχή, στα ύδατα των Κομορών και δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ε, λόγος να επιμένουμε για τις ιδιωτικές συμφωνίες που μπορούν να υπογράψουν οργανώσεις ε, σκαφών ε, ε, που αλεύουν για παράδειγμα υπό σημαία σε ηχελών. Ευχαριστώ κύριος Βαρλέσσα, για να ολοκληρώσει. Ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται προσωρινά από 1η Ιανουαρίου και θα πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσον είμαστε υπέρ ή κατά. Εγώ είμαι υπέρ και προτείνω να υποστηρίξουν και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ. Ah, no, vamos a finalizado este punto, pasamos ahora al punto número 20 Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 20 της ημερήσιας διάταξη, όπως συμφωνήσαμε, ανακοινώσεις του Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστέ. Έχετε τις αποφάσεις εδώ. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Κυρία Ρόντουστ. Sorry. Κύριε Πρόεδρε, χτες το είπα επανειλημμένα. Δεν συμφωνούμε με την με την απόφαση το 2 πιστευουμε ό, άμα πρέπει να φτιαχτεί έκθεση θα πρέπει να ακολουθηθούν οι κανόνες της Επιτροπής μας. Η πολιτική αναλαμβάνει εκείνη η πολιτική ομάδα που έχει τους περισσότερους πόντους εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση ζητούμε την έκθεση αυτή διεκδικούμε την έκθεση αυτή την πληρώνουμε την έκθεση αυτή και θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα σήμερα το πρωί ε, ε, μίλησα με τον Στιούαρτ. Χτες εκείνος πρότεινε να, να γίνει απλώς μία ακρόαση, όχι έκθεση. Να μην γραφτεί έκθεση. Αν είχε αποφασιστεί αυτό θα το δεχόμαστε. Αλλά τώρα δεν αποφασίστηκε αυτό, αποφασίστηκε έκθεση. Αφού πρόκειται για έκθεση θέλουμε να ακολουθηθούν οι κανόνες, την αναλαμβάνουμε εμείς και την πληρώνουμε εμείς. Ευχαριστώ κυρία Ρόντους. Ε, στα πρακτικά φαίνεται αυτό το οποίο συνέβη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αναγράφεται στα πρακτικά, ψηφίσαμε και αποφασίστηκε να αναλάβει την έκθεση η Προεδρία. Αυτό θα πρέπει να επικυρώσει σήμερα η Επιτροπή. Ε, οι συστάσεις των συντονιστών ε, είναι αυτές και αυτό υποβάλλουμε προς ψηφοφορία. Είμαστε υπέρ λοιπόν των αποφάσεων των συντονιστών. Έχετε όλη την κάρτα σας. Κύριε Αρσένη, παρακαλώ. Κύριε Αρσένη. Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ ένα διαδικαστικό θέμα. Βλέπω συναδέλφους που δεν είναι μέλη της Επιτροπής και ποτέ όσοι δεν είναι μέλη δεν μπορούσαν να ψηφίζουν για διαδικαστικά θέματα μέσα στην Επιτροπή. Είναι αγαπητοί συνάδελφοι, τους καλωσορίζω εδώ, αλλά διαδικαστικά είναι καινούριο αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Είστε βετεράνος, τελειώνει η θητεία και θα νόμιζα ότι με κοροϊδεύετε αν δεν ήσασταν βετεράνος. Ε, οι βουλευτέ έχουν δικαίωμα να είναι εδώ, θα ήθελα να μου πει αν είναι νόμιμο η γραμματεία. Ναι, όλοι οι βουλευτέ έχουν δικαίωμα να παραστούν σε οποιαδήποτε επιτροπή και να, να ε, αντικαταστήσουν οποιονδήποτε προβουλευτή. Γίνεται εδώ και πέντε χρόνια και δεν θα αλλάξει σήμερα η διαδικασία γιατί δεν σα αρέσει εσά. Όπως και να έχει, έχετε κάθε ένομο συμφέρον να διαμαρτυρηθείτε, να πείτε ό,τι θέλετε. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λοιπόν, θα ήθελε η Γραμματεία να μου επιβεβαιώσει αν είναι νόμιμο, αν γίνει βάσει των κανόνων αυτό, Πάντα το κριτήριο ήταν επακριβώς το ίδιο. Η Επιτροπή πάντα επιτρέπει να αναπληρώσει οποιοδήποτε βουλευτής, οποιονδήποτε άλλο βουλευτή, είτε είναι τακτικό μέλος είτε όχι της Επιτροπής μας και αυτό το γνωρίζετε. Το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει το αποτέλεσμα είναι άλλο παπά Ευαγγέλωμα. Αλλά δεν θα ψηφίσουμε ό,τι σας αρέσει. Ο κύριος Μιλάνα. Εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς ψηφίζουμε και γιατί πρέπει να ψηφίσουμε. Ποτέ δεν έχουμε επικυρώσει με ψήφο πρακτικά συντονιστών. Να σας εξηγήσω κύριε Μιλάνα. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν γιατί πρέπει να ψηφίσουμε. Θα σας το εξηγήσω πολύ σύντομα. Ποτέ δεν έχουμε ψηφίσει, διότι ποτέ δεν υπήρχαν ενστάσεις ε, στα όσα ε, είχαν προτείνει οι συντονιστές. Το λέω για όσο καιρό ήμουν εγώ πρόεδρος. Και αν υπήρξε οποιαδήποτε ένσταση, επειδή η Επιτροπή είναι αυτή η οποία αποφασίζει και ψηφίζει, αν υπάρχει λοιπόν μια διαφωνία μεταξύ των συντονιστών, το υποβάλλουμε στην Επιτροπή και ψηφίζει η Επιτροπή. Δεν πρόκειται να γίνει περαιτέρω συζήτηση. Η συζήτηση έγινε χθε, έχετε την άποψη των συντονιστών και ψηφίζουμε λοιπόν τις ανακοινώσει για τις ε, αποφάσεις που ελήφθησαν. Υπέρ των αποφάσεων. 11. ¿Votos en contra? Κατά. Έντεκα οκτώ. Για να κάνουμε μια επαλήθευση. Momento, comprobación electrónica. Να κάνουμε λοιπόν μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Ο κύριος Σάλβα δεν έχει κάρτα. Άρχεται η ψηφοφορία.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 Ψήφισαν όλοι, πέρασε τη ψηφοφορία. Δέκα ψήφοι υπέρ, συν μία του κυρίου Σάλβα, κατά οκτώ. Εγκρίνεται λοιπόν η ε, σύσταση των συντονιστών. Διακόπτουμε και θα συνεχίσουμε στις τρεις. Η κυρία Φράγα. Perdón, Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Έχουμε και άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ενημέρωση από τον κύριο Στίβενστον για τα της Task Force. Κύριε Στίβενστον, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ που μου δίνετε το χρόνο να το θέσω το θέμα αυτό πριν τελειώσει η συνεδρίαση. Ησυχία παρακαλώ λέει ο πρόεδρος Silencio, por favor. Λοιπόν, κύριε Στίβενσον, πρόεδρε, δεν θα μπορέσω να είμαι παρόν το απόγευμα, οπότε σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου δίνετε τη δυνατότητα τώρα το πρωί πρωτού να φύγω να σας πω τι έγινε με την Task Force. Όπως ξέρετε, η Task Force δημιουργήθηκε με εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων. Εγώ προείδρευα της προείδρευσα της Task Force για, από πλευράς Κοινοβουλίου για τα πολιετή σχέδια. Πέντε συναντήσεις έγιναν μέχρι τώρα ε, Κοινοβουλίου Κομισιών Συμβουλίου και πριν από τη, τα Χριστούγεννα α, συμφωνήσαμε για για τα μεμονωμένα από και τα πελαγικά είδη είχα, καταφέραμε δηλαδή να συμφωνήσουμε τι θα κάνουμε με τα πολυετή σχέδια για μεμονωμένα ε, αποθέματα, αποθεματα single stocks και υπήρξε λοιπόν συμφωνία και γι' αυτό η Κορεπέρ ε, μετά το Συμβούλιο δηλαδή είπε πολύ ωραία ας αρχής Κομισιόν να φτιάχνει αυτά τα πολιετή σχέδια για τα μεμονωμένα αποθέματα. Τώρα η, στην ελληνική ο ελληνική προεδρία ξεκίνησε, ξεκινάει η δεύτερη φάση αν θέλετε για τις, τη μεικτή αλία, πολλαπλά είδη πολλαπλά αποθέματα. Φαντάζεστε λοιπόν ότι εδώ θα υπάρξουν προβλήματα. Ξεκινήσαμε με προφορική παρουσίαση στα γραφεία του Συμβουλίου. Ο Ερνέστο Πένιας είπε ωραία βασιστούμε στη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε για τα μεμονωμένα θέματα και ας αρχίσουμε λίγο λίγο σταδιακά ας πάρουμε το παρά, παράδειγμα μιας απλής μικτής αλίας όπου κυρίαρχα είναι δύο αποθέματα. Ας πούμε γλώσσα και πλάτακας Και στα πλαίσια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής προσπαθεί κανείς να εξισορροπήσει ας πούμε ένα είδος το οποίο είναι είναι μεγάλο σε ποσότητα, υπάρχει αυθονία σε σχέση με ένα άλλο όπου ε, υπήρξε υπερεκμετάλλευση γι' αυτό δεν έχουμε μεγάλο απόθεμα αυτή είναι η ισορροπία προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε βεβαίως όταν ψαρεύει κανείς για τη γλώσσα και τον πλάτα αλλιεύει και άλλα και άλλους ηχθείς και άλλα είδη. Αυτά δεν πολύ λαμβάνονται υπόψη στο πρώτο παράδειγμα αυτό που κάνουμε με τα δύο είδη. Ε. Βέβαια αν η αλία που κάνει κανείς ε, επαφίεται, βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, το υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, τι γίνεται με τις απορρίψεις, Ας πούμε, ε, εξαντλήσατε την ποσόστοσή σας για ένα είδος και ξαφνικά εμφανίζονται κάποιοι, μια μικρή ποσότητα ηχθείων αυτού του είδους. Τι γίνεται. Τέλο πάντων, αυτά θα τα δούμε, θα τα πούμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το Μάρτιο ε, που θα γίνει μια πρώτη συνάντηση και θα πρέπει να ε, υπάρξει συμφωνία γιατί μην ξεχνάτε ότι τον Απρίλιο, 17 Απριλίου διακόπτει τις εργασίες του το Κοινοβούλιο ενώπιση των εκλογών. Τώρα, ο Υπουργός Αλίας της Ελλάδας χτες είπε ότι αναγνωρίζει τη σημασία των πολιετών σχεδίων. Θεωρεί ότι είναι αναπόσπαστο μέρος της ε, κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Προσπαθούμε λοιπόν να, να δουλέψουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα γίνεται μια συνάντηση τη, τη βδομάδα γίνεται εδώ στις Βρυξέλλες γιατί δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει εκπρόσωπο στο Στρασβούργο προσπαθούμε λοιπόν να επιταλέ, να κάνουμε κάτι τι να προχωρήσουμε τα πράγματα κατά πόσο θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή όχι δεν ξέρω αλλά ευχαριστώ για την υποστήριξή σας Ευχαριστούμε κύριε Στίβενσον και κυρία Φράγα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα στον κύριο Στίβενσον όσον αφορά τις συμφωνίες για την αλληλεία ενός είδου, που είναι οι πιο απλές είναι τη διαφορά απόψεων που υπήρχε μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νομική βάση και θα ήθελα να ξέρω πώς λύθηκε και το θέμα αυτό για την αλληλεία ε, ε, ενός είδους για το Harvest Control Rule. Υπήρχε σαφής διαφορά εκεί μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούσε ότι ο Harvest Control Rule και ο κανόνας αυτός δηλαδή ήταν αρμοδιότητα συναπόφασης, ενώ το Συμβούλιο ανέκαθεν θεωρούσε ότι είναι θέμα το οποίο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Εγώ όταν ε, το άφησα το θέμα αυτό, είχε γίνει μια αντιπρόταση στο Συμβούλιο και έλεγε ότι υπάρχει ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο όριο σε αυτόν τον κανόνα του Harvest Control και αυτός λαμβάνεται υπόψη για την επιστημονική αξιολόγηση ώστε να πληρούνται οι στόχοι που ε, καθορίζονται σε αυτό το τομέα. μέγιστη βιώσιμη απόδοση, MSY σε αυτή την περίπτωση, σε κάποια άλλη περίπτωση ήταν κάποια άλλα. Το θέμα είναι λοιπόν να καθοριστούν τα τάκ και οι ποσοστώσεις μεταξύ αυτού του ελαχίστου και μεγίστου ορίου. Και θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς συνέβη με αυτό. Διότι για μένα η όλη ουσία της συζήτησης ε, ε, που κάνουμε για τη νομική βάση για το Συμβούλιο ήταν ακριβώς αυτός ο κανόνας, το harvest control. Ε, να μην αφήνουμε το Συμβούλιο να κάνει ό,τι του καπνίσει όταν καθορίζονται και ποσοστώσεις. Και θα ήθελα να ξέρω τι έγινε με το Συμβούλιο, πώς το συμφωνήσατε αυτό, διότι μας είπατε ήδη για τα σχέδια διαχείρισης, ε, για συγκεκριμένα είδη. Ε, επομένως έχει ήδη συμφωνηθεί τι γίνεται. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιος άλλος πριν απαντήσει. Ο κύριος Ντέιβις είχε, είχε ζητήσει το λόγο. Question, uh, to... Ήθελα απλώς να πω πόσο χαίρομαι που η ελληνική προεδρία επεξεργάζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επικύρωση αυτής της συμφωνίας γιατί ο κάποιος πολιετής σχεδιασμός της είναι πάντα ζωτικό θέμα. Φοβόμουν ότι το Συμβούλιο μπορεί να έβρισκε τρόπους καθυστέρησης. Αλλά ο Στουαρ Στίβενσον μας είπε ότι το Συμβούλιο τώρα θέλει να λύσει αυτό το θέμα και να προχωρήσουμε. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Yeah, ναι, για να ακολουθήσω λίγο σε αυτά που είπε ο Χρήστος Ντέιβις. Το Συμβούλιο ήδη από τη Λιθουανική Προεδρία μας εξέπληξε γιατί όλοι εξεπλάγησαν από την πρωτοβουλία του να συνεργαστούν τα τρία όργανα σχεδόν σαν τριμερής διάλογος και δείξαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε. Και λόγω αυτού η ελληνική προεδρία είναι πολύ θετικά διατεθειμένη για όλη αυτή τη διαδικασία. Η δε Κάρμεν Φράγα έθεσε το κύριο πρόβλημα, δηλαδή καταφέραμε μέχρι τώρα να πετύχουμε πρόοδο σε αποθέματα ενός είδους αποφεύγοντας να συζητήσουμε το 42.2 και το 42.3. Έτσι το παρακάμψαμε, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αποφεύγουμε αυτή τη συζήτηση. Και μας είπε τις προάλλες ο Πένιας ότι δεν θα κάνουν συστάσεις γιατί θα το συναποφασίσουν οι δύο νομοθέτες. Και εδώ είναι ο κόμπος. Είναι ακόμη εκκρεμές το θέμα στο δικαστήριο, εκκρεμή. Είχαμε πει ότι δεν θα αποδυναμώσουμε τα επιχειρήματά μας, αλλά για να σας πω λίγο νομικά τι συμβαίνει, με την άδεια του Προέδρου θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την νομική υπηρεσία να μας κάνει μια εξήγηση. Ναι, η νομική υπηρεσία. Μπορείτε να μας ενημερώσετε. Ε, yes, with great pleasure, Mr. Chairman. So, actually, what the, the... κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση τώρα είναι ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να κυρωθεί ε, το πολιετές σχέδιο για το γάδο του 2014 και σε αυτή την περίπτωση εμείς ισχυριζόμαστε ότι έπρεπε να εγκριθεί με συναπόφαση βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 2 διότι άπτεται των κανόνων που καθορίζουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα, τα τάξ σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίω σε περιπτώσεις οι οποίες δεν υπάρχουν επαρκή ε, ή υπάρχουν λυπή επιστημονικά στοιχεία. Αυτή είναι η ουσία ε, του λεγόμενου Harvest Control Rule. Και η διαδικασία αυτή δυστυχώς θα καθυστερήσει κι άλλο, διότι προς το παρόν βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της αρχικής διαδικασίας, δηλαδή ε, γράφουμε τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου ε, στις δηλώσεις και παρεμβάσεις κάποιων χωρών ε, μελών που παρουσίασαν παρουσια, ε, παρατηρήσεις για να υποστηρίξουν το Συμβούλιο και μετά από αυτό το στάδιο θα χρειαστούν πάρα πολλοί μήνες πριν υπάρξει ακρόαση από το δικαστήριο και πάλι και μετά και άλλοι μήνες μπορεί ε, να περάσουν μέχρι να έχουμε την άποψη και του εισαγγελέα αλλά και την τελική απόφαση. Μέχρι να τη λησιδικήσει δηλαδή απόφαση μάλλον θα περάσει ένας χρόνος τουλάχιστον. Αυτό όμως που έχει σημασία και που είπε και ο κύριος Στίβενσον είναι ότι τελικά το δικαστήριο είναι το μόνο το οποίο μπορεί να ερμηνεύσει οριστικά τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη συνθήκη. Επομένως, όταν θα υπάρξει τελεσίδικη απόφαση θα ισχύει για όλες τις μελλοντικέ περιπτώσεις και θα καθορίζει ε, σε αυτή τη διαδικασία ποιο τμήμα των πολιετών ε, σχεδίων θα εγκρίνονται και φυσικά η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι και η θέση που υπερασπιζόμαστε στο δικαστήριο είναι ότι όλα τα πολιετή ε, σχέδια διαχείρισης θα πρέπει να αποφασίζονται ως συναπόφαση γιατί θεωρούνται ως σύνολο. Πριν υπάρξει όμως ε, τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι και τίποτα δεν απαγορεύει εντωμεταξύ στο να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις και να συμφωνήσουμε μια κοινή προσέγγιση για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε ε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Από νομική σκοπιά, αυτό το οποίο αντιλήφθηκα εγώ στη συνεδριάση της Task Force ε, στην οποία, ε, στις οποίες ήμουν παρόν, είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, τα θεσμικά όργανα ακολουθούν άλλη προσέγγιση. Δεν συζητούν πλέον αυτούς τους κανόνες ε, του harvest control που ε, υπήρχαν στα προηγούμενα σχέδια, αλλά εξετάζουν ποιες παράμετροι θα ληφθούν υπόψη για να καθοριστούν τα τάκ και η αλληλευτική προσπάθεια στο μέλλον. όχι απαραίτητα λοιπόν υπό τη μορφή κανόνα harvest control όπως το γνωρίζουμε, αλλά όπως ε, έχουν συζητηθεί μέσω επιστημονικών ε, ε, ορίων ή κάτι αντίστοιχο. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία είναι ότι οποιοδήποτε μηχανισμός θα καθορίζει στο τέλος πώς αποφασίζονται οι αλευτικές δυνατότητες θα πρέπει, ε, τουλάχιστον όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τη συνθήκη, θα πρέπει να λαμβάνεται σε συναπόφαση. Τώρα, αν θα τον λέμε harvest control rule ή καθορισμό παραμέτρων που θα προκαθορίζουν εντός ποιού φάσματος θα εμπίπτουν τα τάκη ποσοστώσεις, δεν έχει σημασία. Η συζήτηση αυτή όμως είναι αυτή τη στιγμή στα σπάργανα και δεν ξέρουμε πολύ περισσότερο όταν θα περατωθεί. Το βασικό μήνυμα όμως το οποίο θα ήθελα να σας διαβιβάσω είναι ότι εάν δεν υπάρξει απόφαση του δικαστηρίου δεν θα μπορούμε να γνωρίζουμε ε, σίγουρα και η απόφαση αυτή υπορτερεί ακόμα και σε οποιαδήποτε διεθνή διαπραγμάτευση. Γιατί ακόμα και αν ε, λάβει τη μορφή μιας ε, διοργανικής συμφωνίας, κάτι το οποίο δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, όπως λέει ο κανονισμός στο άρθρο 157, ακόμα και αυτό δεν θα είναι νομικά δεσμευτικό. Δεν μπορεί να πάει... Δεν μπορεί, συγγνώμη, να θεωρηθεί ότι υπερτερεί τη απόφαση του δικαστηρίου. Πριν όμω έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου, δεν θα ξέρουμε ακριβώ τι θα ισχύει. Ευχαριστώ. Bien, muchas gracias al servicio jurídico. ¿Hay alguna otra... Ευχαριστούμε την νομική υπηρεσία. Άλλος κανείς? Όχι, ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Στίβενσον για την ενημέρωση και τώρα λοιπόν διακόπτεται η συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε στις 3 με την ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Δαμανάκη. Τα λέμε το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.